Tisztelt Ház, kedves képviselőtársaim! Megkezdődnek a szavazás. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι επεξηγήσεις ψήφου τώρα για την έκθεση Άλβαρο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ανδρικίνε. Για ένα λεπτό. In favor of the agreement between the... Υπερψήφισα τη συμφωνία Πολιτειών και Ευρωπαϊκή Ένωση, για την επεξεργασία και διαβίβαση χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει απειλή για την ίδια την ασφάλειά μα και για την ασφάλεια των εταίρων μα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Να σα θυμίσω. Δεν χρειάζεται να σα θυμίσω τι θερμοκρατικέ επιθέσει που δεχτήκαμε και έλαβαν χώρα στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας είναι στρατηγικός εταίρος όχι μόνο στην περιοχή της παγκόσμιας ασφάλειας αλλά και από την άποψη την οικονομική και από κάθε άποψη. Η στρατηγική αυτή εταιρική σχέση εκφράστηκε από τον πρόεδρο Biden πριν από λίγους μήνες. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε λοιπόν ότι συνενέσαμε σε μια συμφωνία που είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη οποιασδήποτε τρομοκρατικής δραστηριότητας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά γιατί το Κοινοβούλιο επέφερε σοβαρές διευκρινήσεις στην έκθεση αυτή που θα πρέπει να ληφθούν, στη συμφωνία αυτή που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κύριος Μπάτεν σε ένα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολλοί λόγοι να καταψηφίσει κανείς αυτή την ε, έκθεση και συμφωνία, αλλά δύο πράγματα θέλω να καλύψω σε 60 δευτερόλεπτα. Ότι βεβαίω πρέπει να καταπολεμήσουμε τη δημοκρατία, αλλά αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ώστε οι κυβερνήσεις να κατασκοπεύουν τους πολίτες τους. Τα απόρριτα στοιχεία που αφορά η συμφωνία αυτή ανήκουν στον κάθε πολίτη, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο ή και σε καμία περίπτωση τι Πολιτείε ή το Εθνικό Κράτο. Κάθε τέτοια συμφωνία πρέπει να συνάπτεται μεταξύ των κυρίαρχων εθνικών κρατών που μπορούν και να είναι υπόλογα προ του πολίτε του μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών. Εδώ βεβαίω έχει υπογραφεί συμφωνία, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε για καμία βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ θα τον τιμήσουν. Ω προ τον Βρετανικό νόμο για την προστασία των δεδομένων, απαγορεύεται η διαβίβαση πληροφοριών χωρίς, με, τρίτα μέρη χωρί την συνένεση του ενδιαφερομένου. Και η Βρετανική κυβέρνηση έχει ρήτρα εξαίρεση από την. Ε, ε, συμφωνία αυτή. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι θα αντιταχθούν στην κατασκοπία και θα ακολουθήσουν τη δική μου τη στάση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάσμαρεκ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση του κύριου Αλβάρο γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πραγματικό εργαλείο, ουσιαστικό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και παράγον σημαντικό σε αυτό, είναι η προληπτική δράση, δηλαδή ο έλεγχος των οικονομικών, των κονδυλίων που τρέφουν την τρομοκρατία. Εάν μπορέσουμε αυτά να τα ελέγξουμε, τότε θα υποχρεώσουμε και την τρομοκρατία σε έναν βέβαιο θάνατο. Και χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για το σκοπό αυτό όλοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάκουλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα και εγώ την έκθεση Όλβαρο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού την τρομοκρατία. Έχουμε κοινέ αξίες και με τους εταίρους μας πρέπει να αγωνιστούμε για να τις διαφυλάξουμε. Είναι σαφές ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να τη φυλάσετε και στον αγώνα κατά την τρομοκρατία και πιστεύω ότι θέσαμε τα όρια της διαφύλαξης ε, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που δεν μπορούμε ούτε για λόγους καταπολέμησης τρομοκρατίας να υπερβούμε. Νομίζω ότι μπορούμε με τον τρόπο αυτό να είμαστε βέβαιοι ότι θα φέρουμε την ειρήνη στον κόσμο καταπολεμώντας την τρομοκρατία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Χάναν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντοτε είναι ευαίσθητη η ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών των, πολιών, των πολιτών και τη ασφάλεια. Και πολλέ φορέ από τι επιθέσει τη 11η Σεπτεμβρίου πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει τη σωστή ισορροπία. Και αυτό γιατί υπάρχει μια λανθασμένη εξίσωση στην πολιτική. Δηλαδή, οι πολιτικοί θύνοντε πιστεύουν ότι οι δράσει του πρέπει να είναι αναλογικέ σε σχέση με την οργή του κοινού και όχι σε σχέση με την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε και να εντοπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Και το δικό μα κοινοβούλιο έχει κάνει το λάθο αυτό, αλλά και εθνικά κοινοβούλια και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε πετύχει τη σωστή ισορροπία. Διότι έχουμε σκεφτεί αρκετά, έχουμε λάβει υπόψη όλα τα ενδιαφέροντα όλων των μερών και ιδίω οι δυνάμει καταστολή ε, διεθνώ που καταπολεμούν ε, σε κοινή συνεργασία αποτελεσματικά την τρομοκρατία έχουν λάβει υπόψη επαρκώς και τις ανάγκες ε, ελευθερίας των ε, πολιτών. Και αυτό είναι βεβαίω και ο στόχο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί αυτό να επαφείται μόνο στα κράτη-μέλη. Πολύ σωστά λοιπόν επετέφθη η συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση, έκθεση Μπροκ. Πρώτο ομιλητή, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ καταψήφισα την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διότι θεωρώ ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να εξασθεί στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Οι αλλαγές λοιπόν που έχει υποστεί αυτή η πολιτική υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, προσφέρουν περισσότερους σπόρους για την ενίσχυση των εξοπλισμών στην Ευρώπη και με τη συνθήκη αυτή τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρώπης που είναι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις ταυτόχρονα, θα έχουν ε, περισσότερη ευχέρεια για ανάληψη και εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών. Είναι αναμφίβολα ε, δεδομένο ότι στο μέλλον θα μπορούν τα κράτη αυτά τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλαμβάνουν δραστηριότητες στρατιωτικές στα τρίτα κράτη, οποτεδήποτε θεωρούν ότι το οικονομικό του συμφέρον το επιτάσσει. Και όπως άλλωστε κάνουν οι ΗΠΑ Πολιτείες. Προβάλλουν δηλαδή και προωθούν τις οικονομικές αξίες του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού, πράγμα το οποίο με να με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εγώ στήριξα την έκθεση του κυρίου Μπροκ, γιατί η κοινή θέση του Ευρωκοινοβουλίου έχει αξιοποιήσει πλήρως τις νέες ευκαιρίες που η συνθήκη της Λισαβόνας μας προσφέρει. Στηρίζω ιδιαίτερως την πολιτική και οικονομική εποπτεία του Ευρωκοινοβουλίου ως προς τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνένεση της είπα εκπροσώπου να, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ειδικό εκπρόσωπο στην έδρα αυτή τη υπηρεσία είναι πολύ σημαντική. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει και απαραίτητη γεωγραφική ισορροπία μέσα σε αυτή την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, με εκπροσώπου και από τα 27 κράτη-μέλη. Η διαδικασία αυτή μόλις έχει ξεκινήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό η αναθεώρηση του 2013 να λάβει υπόψη και το θέμα αυτό της ίσης γεωγραφικής εκπροσώπησης των κρατών μελών. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Αντρικένε για ένα λεπτό. Yes, I missed... Μάλλον όμως ξέχασα Ο κύριος Αντωνιούτσι, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα είναι ένα βήμα καθοριστικής σημασίας, ε, ιστορικής μάλιστα, για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι εδώ υπογραμμίζουμε τη σημασία μεγαλύτερη, την ανάγκη μεγαλύτερης συνέπειας στη δράση της υπηρεσία αυτής και να υπάρξει συντονισμό μεταξύ των ε, δημοκρατικών υπηρεσιών των κατομελών και της ΙΑΗ και της ε, εξωτερικής ε, υπηρεσίας αυτής. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μακροπρόθεσμα δεν θα δημιουργηθούν κάποιες αντιφάσεις με τα γεωγραφικά, στατηγικά και πολιτιστικά συμπέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και να τα φροντίσουμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή, η επόμενη ομιλήτρια, μάλλον η κυρία Ντούτσεν, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την έκθεση. Και τη μερική εδώ παρόντες ε, είναι εκστασιασμένοι με την υπέροχη αυτή υποτίθεται έκθεση και τη δημιουργία της, της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο αισθάνεται μεγάλη απογοήτευση και ε, ενόχληση από το γεγονός ότι διαβρώνεται διαρκώς η εθνική του κυριαρχία και επικρατεί ο φόβος ότι μπορούμε τελικά να βρεθούμε ε, υπόδουλοι σε κάποιον ο οποίος δεν είναι άμεσα εκλεγμένος από τον Βρετανικό λαό. Μας υπόσχονται τώρα ότι αυτή η υπηρεσία θα έχει μεγάλη επιτυχία, μεγάλη συμβολή στην ε, επιτυχή ε, ανάληψη ρόλου παγκοσμίου στο διεθνέ σκηνικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν ξεχνάει ότι χάνονται, ότι γίνονται περικοπές από τον εθνικό προϋπολογισμό 40% από τις κρατικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα ε, μας υπόσχονται δαπάνες 900 εκατομμυρίων ευρώ που δεν τα χρειαζόμαστε ούτε τα θέλουμε από την υπηρεσία αυτό. Είμαστε λοιπόν όλοι κατά αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κόρχολα έχει το λόγο. Kiitos arvoisa puhemies. Ε, unionin ulkosuhdehallinnon perustamista koskevassa äänestyksessä kannatin muutosesityksiä, jotka korostavat kansallisten parlamenttien mukaan. Ευχαριστώ πολύ η επαλήθευση των δραστηριοτήτων αυτών πρέπει οπωσδήποτε να ε, ανήκει στα, κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε την ε, διαφάνεια και τη λογοδοσία αυτής της υπηρεσίας και ιδιαίτερα ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί το δυσάρεστο φαινόμενο της υποχρηματοδότησης των ΗΕ και στην υπηρεσία αυτή. και πιστεύω ότι θα τηρηθούν οι διεθνείς κανόνες. Ευχαριστώ, κυρία Βάιντερα. Πρόεδρε, Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, θα βοηθήσει την βελτίωση και πιο αποτελεσματική οργάνωση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ένας παράγων στη διεθνή σκηνή. Πρέπει ωστόσο να ρυθμιστούν επιμέρους ζητήματα, διαφορετικά θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η υπηρεσία. Πρέπει να καταστεί προτεραιότητα η γεωγραφική εκπροσώπηση, ισοδύναμη γεωγραφική ε, εκπροσώπηση, πρέπει να υπάρχουν βασικές υπηρεσίες, πρέπει επαγγελματισμός και ισόρροπη δράση να είναι οι επιλογές από την πρώτη μέρα ανάληψης δραστηριοτήτων αυτές της υπηρεσίας. Η συμβιβασμοί και η αναλογική ε, ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας νομίζω ότι μπορούν να οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριο Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι σήμερα. Έχουμε φτάσει σε μια απόφαση που θα καταφέρουμε, με την οποία θα καταφέρουμε να επιταχύνουμε την ε, ίδρυση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όμως είναι πολλά αυτό που ακόμα επομένει να γίνουν. Η εμπορική μας πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά δεν μπορούν να είναι θέματα που εξετάζονται ανεξάρτητα από την εξωτερική πολιτική. Οι οικονομίες μας πλέον είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και έχουν άμεση σχέση και με την εξωτερική πολιτική. Έπειτα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, να βεβαιωθούμε ότι έχει τον απαραίτητο έλεγχο και τις δυνατότητες εποπτείας ε, στο κοινοβούλιο ίσως αυτό και ίσως θα έπρεπε να είναι ένας ξεχωριστός φορέας αυτός που θα δημιουργηθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που να συνεργάζεται με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες. Βέβαια τέτοιου είδους ε, αποτελέσματα για να επιτευχθούν χρειάζονται χρόνια πολλές φορές. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε απόψη αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις συνθήκες της Λισαβόνας, όμως πρέπει να πω ότι έχω και κάποιες αμφιβολίες για την όλη αυτή προσπάθεια. Εδώ δημιουργούμε ένα ολόκληρο διοικητικό οικοδόμημα και λέμε ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ουδετερότητα, πράγμα που δεν είναι αναγκαίο ότι θα συμβεί. Πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για τους Ευρωπαίους. Και έχουμε το αξίωμα του είπατε εκπροσώπου, ξέρουμε ότι θα κοστίσει. Γι' αυτό λοιπόν να μην ξεκινάμε με ψέματα. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερο είναι ότι τα μεγάλα κράτη-μέλη έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος μέσα στις δομές αυτές πρέπει να έχουμε καλύτερη εξισορρόπηση και εκπροσώπηση και πρέπει να έχουμε και εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου για να εκπροσωπούνται όλα τα κράτη ισοδύναμα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ο κύριος ε, Μάρτιν έχει το λόγο. Πρόεδρε, χαίρομαι για την ψηφοφορία, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά τώρα που έγινε αυτή, καλό θα είναι να αφήσουμε τις δομές και τις διαδικασίες κατά μέρο και να κοιτάξουμε τι δουλειά θα κάνει αυτή η υπηρεσία. Η κάθε Άστον πρέπει να γνωρίζει ότι έχει στο πλευρό της μια ομάδα η οποία τις ευρωπαϊκές αξίες τις θέτει στην, στην κύρια προτεραιότητα με πάνω απάνω τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει υπηρεσία ειδική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να αναλάβει και κάποιος ε, ως μέλος του επιτελείου της το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων για να τα παρακολουθεί εκ του σύνεγγης. Όταν λοιπόν έχουμε χώρες, με πρώτη-πρώτη την Κίνα, για τις, οποίες, για τις οποίες χώρες ο υποτιθέμενος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ε, μηδενική σημασία, καλό θα είναι να αρχίσουμε, να υποστηρίζουμε και να αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάναν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εδώ κάτι μου φαίνεται σχεδόν συγκινητικό με τι συζητήσει μα αυτέ και το πώ θα δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Λε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε μια, ένα πλήρη εξοπλισμό με διπλωματικέ υπηρεσίε. Διότι οποιαδήποτε τρίτη ε, χώρα θα έχει μια Ευρωπαϊκή Πρεσβεία η οποία θα στεγάζει προφανώς ε, προσωπίες των ε, ευρωπαϊκών κρατών. Εδώ φαίνεται να έχουμε ήδη πιέσει για τους μισθούς της είπα εκπροσώπου που είναι 20 πλάσια από όσα ισχύουν για την αντίστοιχη θέση στο εθνικό κράτος, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε να κάνουμε Κάτι τελείω ξεχωριστό σε σχέση με το τι κάνουν τώρα τα διπλωμα... οι διπλωματικέ υπηρεσίε στην ε, Ευρωπαϊκή... τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ταϊβάν, στην Κούβα, με την Χαμά, ε, στο Ισραήλ. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε την μεγαλύτερη, την πέμπτη οικονομική δύναμη στον κόσμο και θα πρέπει να κάνουμε τη δική μα ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Σα ευχαριστώ. Και εν τέλει, η κυρία Γκρέσλε για ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την έκθεση Μπροκ. Γιατί αποδυναμώνεται σημαντικά η δομή αυτής της υπηρεσίας ε, κατά τρόπο πολύ ανησυχητικό. Επίσης, οι πρεσβείες θα αρχίσουν τώρα να, διαχειρώνονται, να διαχειρίζονται κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Και επίσης εδώ το Κοινοβούλιο έχει εμπλακεί σε ένα κανονισμό του Συμβουλίου με μια διαδικασία που de facto ήταν συναπόφαση, αλλά όπου επιτρέψαμε δυστυχώς στο Συμβούλιο να ε, κρατήσει, να παρακρατήσει μεγάλο μέρος των εξουσιών που ανήκαν σε εμάς. Δυστυχώς. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω πώς πρόκειται να συνεργαστούμε μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί στην προηγούμενη θετία εγκρίναμε μία μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου, την οποία τώρα καταπατούμε ήδη με αποφάση και σύμπραξη του Προεδρείου και τη δέσκεψη των Προέδρων. Τι να την κάνουμε λοιπόν, τη μεταρρύθμιση, εάν ήδη στου πρώτου μήνε τη λειτουργία τη νέα θητεία την έχουμε καταπατήσει σε τέτοιο βαθμό. Ευχαριστούμε. Οι εξηγήσει ψήφων θα συνεχιστούν με την πρόταση ψηφίσματο για το κοσυφοπαίδιο. Δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος της δικής μου ομάδας για το κοσυφοπαίδιο, διότι δεν είχα άλλη επιλογή. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ουσίας στην έκθεση αυτή, τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο. Θεωρώ ότι το κοσμοπέδιο πρέπει να έχει μια βιώσιμη δημοκρατία, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, μια κοινωνία όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ναι, λοιπόν, και εγώ επιθυμώ να υπάρχει σταθερότητα στο και δημοκρατία στο Κωσυφοπαίδιο, αλλά προέρχομαι από μια χώρα η οποία δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της, ε, του Κωσυφοπαιδίου και ως εκ τούτου η ε, πληθώρα αναφορών στο κείμενο αυτό τη, του Κωσυφοπαιδίου ως ανεξάρτητου κράτους για μένα είναι απαράδεκτη. Και δεν ελέγχεται δυστυχώ υπόψη το γεγονό ότι δεν έχει αναγνωριστεί από όλε τι χώρε η ανεξαρτησία τη χώρα αυτής του κοσφοπεδίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρέντα και τώρα η κυρία Ντεορκίζα. Πρόεδρε, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, κανένα ε, Ισπανός σοσιαλιστής δεν ψήφισε για να δεχτεί ή να απορρίψει ρητός την ε, ε, ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Εδώ λοιπόν καταψηφίσαμε ακριβώ το ψήφισμα αυτό για να δείξουμε ε, τι αντιρρήσει μα. Εδώ κλήθηκαν τα κράτη-μέλη να ε, στηρίξουν ε, την περιοχή αυτή. Εμείς θελήσαμε όμως να εκδηλώσουμε την, αντί, την αντίρρησή μας σε σχέση με την έλλειψη Στήριξη από τον ΟΗΕ ή από κάποια άλλη διεθνή απόφαση που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Και στα Βαλκάνια οι κάτοικοι όπως φάνηκε από την σύνοδο που οργάνωσε η Ισπανία τον Ιούνιο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως προς τις κέντρες ανάγκες. Τους ευχαριστούμε κυρία Αντρικένα για ένα λεπτό. Ω προ το ψήφισμα αυτό ήθελα να σχολιάσω ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το πολύ σημαντικό θέμα του μέλλοντο του, Κωσο, στο Κωσυφοπέδιο έχουμε το τελευταίο τμήμα του πολύ πολύπλοκου και ευαίσθητου πολιτικού πάζλ των Βαλκανίων. Θα πρέπει λοιπόν εδώ η διαδικασία να ολοκληρωθεί με τρόπο αρμονικό και ειρηνικό. Η ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου έχει αναγνωριστεί από 69 χώρε, μεταξύ των οποίων 22 κατημέλη μελη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να σημειώσουμε ότι με την ε, προοπτική προσχώρηση τη χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τι Βαλκανικέ χώρε να προβούν στι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να επιστρέψουν στην αρχική του σταθερότητα. Αυτό το κοσμοπέδιο δεν είναι βεβαίω εξαίρεση σε αυτή τη διαδικασία. Το κοσμοπέδιο θα έπρεπε να μπορεί να έρθει στην Ευρώπη για να πετύχει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνευση. Και αυτό θα βοηθήσει την ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα και το κοσμοπέδιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ την κυρία Λούνατσεκ για την πολύ καλή συνεργασία εκ μέρου του ΕΛΚ. Το κείμενο το οποίο υιοθετήσαμε σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε στην Επιτροπή. Και εξασφαλίσαμε ότι δεν είναι θέμα επιλογής το κοσφοπέδιο. Τα πέντε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος πρέπει να το πράξουν. Και αυτό είναι λογικό, διότι το 2005 και το 2007 με πλειοψηφία των τριών τετάρτων το Κοινοβούλιο αν, εκάλεσε, ε, ε απεύθυνε έκλεισε για την ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου. Και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν διαπραγματευόμαστε και πάλι το καθεστώς της χώρας. Ο κύριος Πραντσιέρη, τον οποίον κατά τα άλλα εκτιμώ, δηλώνει σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι γίνεται επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος του Κοσμοπέδιου, Πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε σύγχυση και πολλά περισσότερα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το κοσφοπέδιο να μπει μέσα στη διαδικασία του screening, δηλαδή στην προεταξιακή στρατηγική. Και τώρα, τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Χάναν. Κύριε Πρόεδρε, από τις πρώτες ημέρες των συνθηκών των Παρισιών και της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε βάλει τον υπερεθνικό χαρακτήρα πάνω από τον οποιαδήποτε εθνική δημοκρατία. Εδώ λοιπόν είδαμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις της τεχνητής ένωσης ενός πολυεθνικού κράτους. Ακούσαμε Εάν ε, θα... Ακούσαμε τι έγινε με το δημοψήφισμα στο Κοσμοπέδιο και ξέρουμε ότι το 90% του πληθυσμού υπερψήφιζε την ανεξαρτησία. Ξέρουμε όμως τι γίνεται και με τις μειονότητες στην χώρα αυτή και σε όλα τα σύνορα. Επίσης, οι ε, Σέρβοι έκλεισαν τα σύνορά τους προς το Κοσμοπέδιο και τελικά έχουν αποκλειστεί οι πολίτες της μιας και της άλλης χώρας από τις δύο πλευρές των συνόρων. Έτσι λοιπόν αποδεικνύουν τα πολυεθνικά κράτη ότι δεν μπορούν τεχνητά να κρατάμε μαζί διαφορετικές εθνότητες. Αυτό το αποδεικνύουν το παράδειγμα της, της πρώην Γεκουσλαβίας, της Σοβιετικής Ένωσης και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν η κυριαρχία του κατεκάτω σε αυτοκυριαρχία του να αναγνωρίζεται. Ευχαριστούμε. Ε, ακολουθούν οι επεξηγήσει ψήφου για την Αλβανία και παρακαλώ την κυρία Ανδρική να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό. Θεωρώ ότι για άλλη μια φορά θα πρέπει να επαναλάβουμε την υποστήριξή μας προς τις φιλοδοξίες για ευρωπαϊκή ενοποίηση των κρατών της Βαλκανικής μέσα από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η Αλβανία είναι, είναι μια χώρα η οποία έχει ε, κάνει σημαντικές πρόοδους ε, στις μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια χώρα που χρειάζεται ακόμη πολλές πρόοδους να υλοποιήσει για να προσεγγίσει τα προδιαγραφέ τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια ένταξη. Πολλέ περισσότερε προσπάθειε χρειάζονται για την εδραίωση τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου και την εξασφάλιση μια αηφόρου ανάπτυξη στη χώρα. Η δημοκρατική κρίση τον Ιούνιο του 2009 μετά τι ε, εθνικέ εκλογέ ήταν λυπηρό γεγονό και πρέπει να καταστήσουμε ε, σαφέ προ του Αλβανού εταίρου μα ότι η σαφή εκπροσώπηση των θεσμών και ιδιαίτερω του, του Κοινοβουλίου που είναι το πιο σημαντικό αποτελεί την σπονδυλική στήλη ενό δημοκρατικού συστήματο και βέβαια ένα βασικό κριτήριο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Μπεν Πόστολ, είναι επόμενο ομιλητή. Οι πρώην κομμουνιστέ και σοσιαλιστέ τώρα τη Αλβανία προσπαθούν να διαφυλάξουν το καθεστώ που του είναι οικείο. Το γνωρίζουμε αυτό. Δυστυχώ, όμω το ίδιο γίνεται τώρα στη Μακεδονία ίδια προσπάθεια. Προχτές είχαμε τον ε, κύριο Τσεβερκόφσκι εδώ, τον ε, σοσιαλιστή επικεφαλής ε, της αντιπολίτευσης, ο οποίος συνομίλησε σε μυστική συνομιλία με τον κύριο Φιούλα και μάλιστα αυτό αντίθετα με κάθε κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργία του Κοινοβουλίου προέβη και σε δηλώσεις στον τύπο λέγοντας ότι τον, του απέδωσε δίκαιο ο κύριος Επίτροπος ως προς τις θέσεις του στην εσωτερική πολιτική. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένας επίτροπος να δέχεται, να αφήνεται να, τον να καταχρούνται τον... του ονόματός του, να καταχρούνται του ονόματός του κάποιοι για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Η κυβέρνηση της Μακεδονία έχει νομιμοποίηση δημοκρατική, κάνει καταπληκτική δουλειά, φέρνει τη χώρα πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να ασκεί το αντιπολιτευτικό της έργο, αλλά δεν μπορεί να καταχράται του ονόματος και τον... Ε, του θόκου κάποιου ε, αξιωματοχού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε την κατάσταση του Κυργιστάν. Κύριε Αντρικίενα, και πάλι. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που καταδικάζουν τα βία επεισόδια ε, στο Κυργιστάν τον περασμένο μήνα. Είναι πολύ κρίμα που εκατοντάδες στρατιώτες ε, επέλασαν στις δρόμους της πόλης, πυροβολώντας πολίτες και βιτρίνες καταστημάτων και αυτό βάσει κριτηρίων εθνοτικών. Ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για, τους περίπου, για τις οικογένειες των περίπου 300 ε, νεκρών και των 200 τραυματιών που νοσηλεύτηκαν. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να πιέζει τις αρχές της χώρας αυτής, ώστε να έχουν αμερόληπτη, ε, αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για να δουν γιατί προέκυψαν τα δύο αυτά επεισόδια. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βάιντερ. Οι εθνοτικές ε, βιαιότητες, οι διεθνοτικές βιαινότητες στον Ιούνιο ε, ανέτρεψαν ε, τα δεδομένα που γνωρίζαμε. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι τραυματίστηκαν, χιλιάδες ήταν αυτοί που κατέληξαν στα νοσοκομεία και πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλυθούν τα προβλήματα. Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε το Κυργιστάν λοιπόν και για να το βοηθήσουμε θα πρέπει να κοιτάξουμε τους ανθρώπους και όχι την κυβέρνηση. Στις 22 Ιουνίου συναντηθήκαμε μέσω της αντιπροσωπείας μας με τον πρεσβευτή Αζήλοφο, ο οποίος μας είπε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, καμία βιοπραγία και ότι κακός ο τύπος μετέδωσε αυτά που ε, μετέδωσε διότι ήταν ψεύδι. Και όμως Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές, πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα για τους αγωνιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων στο Κυργιστάν. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, πρέπει να συνομιλήσουμε με τα κράτη, ε, τα όμορα του Κυργιστάν, αλλά και με την Κίνα και με την ε, Ρωσία, ε, όσους δηλαδή μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην περιοχή αυτή. καλό θα ήταν να προσκαλέσουμε διεθνείς παρατηρητές και να ζητήσουμε μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα της υπόθεσης αυτής. Ευχαριστούμε. Το επόμενο θέμα τώρα. Ο ιός του AIDS, HIV. Η κυρία Σαμπόρσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μετά από 30 χρόνια ενεργούς πολιτικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις αφρικανικές χώρες, η έκθεση που συζητήσαμε σήμερα διαπιστώνει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από τον ιό HIV έχει αυξηθεί. Το 2008 είχαμε αύξηση 7 εκατομμυρίων ασθενών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν επενέδυσε εκατομμύρια ευρώ για τα προγράμματα περίθαλψης των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει λοιπόν κάποιος λόγος να πιστεύουμε, να σκεφτούμε τι κάνουμε σωστό και τι κάνουμε λάθος αυτή τη στιγμή. Ίσως τελικά η χρήση των προφυλακτικών δεν είναι η μόνη λύση, αλλά η πίστη στη στους συζυγικούς Είναι πολλά αυτά που σήμερα μια γυναίκα μπορεί να πετύχει, έστω και αν ε, υποφέρει από τον ιό αυτό, ε, όπως και να γεννήσει ένα υγιές παιδί σε πολλέ αφρικανικέ χώρε βλέπουμε να μην υπάρχει κατάλληλη πολιτική όμω. Ήταν αναπαγορικά δικαιώματα να μην συνδυάζονται με την υγειονομική αυτή κάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα κατά πολέμησης του ιού αυτού. Και τώρα περνάμε στα όπλα διασποράς. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. προτίμησα την αποχή γιατί η προθεσμία για το άρθρο 2 που αναφέρονται στην ε, Ρουμανία είναι πολύ περιοριστικέ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις σχετικές με τη σύμβαση περί απαγόρευσης ορισμένων ε, συμβατικών όπλων. Και θεωρούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι το κατάλληλο πολυμερές ε, πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συζητηθεί το ζήτημα των όπλων διασποράς. 110 είναι τα κρατη που συμμετέχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εκεί λοιπόν να πρέπει να δοθεί το βάρος. Ευχαριστούμε και τώρα το μέλος της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Είναι αρκετοί οι βουλευτές που έχουν παραμείνει στην αίθουσα. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κολινόφσκι. δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Οπότε, ο κύριος Γιάρ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική είναι μια επιτυχημένη πολιτική και γι' αυτό χάρηκα για την ευρύτερη υποστήριξη τη έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Έχουμε καταρχά σταθερή προμήθεια τροφίμων για τους πολίτες μας, έχουμε την διαφύλαξη της γεωργίας μας και του γεωργικού τομέα και τρίτον έχουμε την προστασία της κλωρίδας και της πανίδας και του περιβάλλοντος μας. Βεβαίως έχουμε τον στόχο της πράσινης ανάπτυξης με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Συμφωνούμε με μια ε, κοινή γεωργική πολιτική ε, εκτεταμένη μια ε, γεωργική πολιτική η οποία διαφυλάσσει όπως, την ορίζει κατά εξαιρετικό τρόπο αυτή η έκθεση. Και ταυτόχρονα η έκθεση υποστηρίζει ένα μοντέλο δύο πυλώνων της κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν τώρα να υποστηρίξουμε την κατάλληλη πρικοδότηση, την κατάλληλη χρηματοδότηση δηλαδή αυτής της κοινωνικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Λάιον γιατί συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς την απέτηση να σχεδιαστεί μια κοινή γεωργική πολιτική που από τη μια να ε, προβλέπει μια ευρεία μεταρρύθμιση τα προσεχή χρόνια και από την άλλη να θέτει πρακτικές προϋποθέσεις και να δίνει λύσεις πρωτοπορίας στις πολυάριθμες υποκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι τα πέντε βασικά στοιχεία που περιγράφονται στην έκθεση, δηλαδή η επισητιστική ασφάλεια, η αηφορία, η γεωργία στην Ευρώπη, η βιοπικιλότητα και η προστασία του περιβάλλοντος, και τέλος, η πράσινη ανάπτυξη είναι άριστα σημεία αφετηρίας ώστε να διασφαλίσουμε μια μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του τι συμβαίνει στο διεθνές προσκήνιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος, η κυρία Κλά. Η έκθεση Λέων για την κοινή γεωργική πολιτική αποτέλεσε μια κοινή έκφραση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σαφής σαφή καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή, κατέγραψε σαφή καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι για την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των συναδέλφων και υποστήριξη στην έκθεση αυτή, κατά την ψηφοφορία, γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η προμήθεια επαρκών τροφίμων και η αηφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του γεωργικού τομέα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τον υποστηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον να εξασφαλίζει την επάρκεια των προμήθεια σε τρόφιμα για του πολίτε τη και ταυτόχρονα έχει μεγάλη ευθύνη και για λόγους περιβαλλοντικούς στην ε, διαφύλαξη αυτών των συνθήκων για τους πολίτες της. Πρέπει όμως να συνεργαστεί με, τον, με τις υπόλοιπε χώρες του κόσμου. Ο γεωργικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει εγγυημένα επαρκή εισοδήματα και σε τελευταία ανάλυση θα μπορούσαμε ίσως να εισαγάγουμε ε, τρόφιμα γεωργικά από άλλες χώρες αλλά με τους όρους στους οποίους εμείς ορίζουμε έτσι ώστε να έχουν και ισότιμο ανταγωνισμό οι γεωργοί μας στους οποίους αξίζουν έπαινοι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σικέσκι. Ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προχωρήσουν ο μηχανισμός ε, παρέμβασης κατά τρόπον ώστε να μην ε, χάσουν τα εισοδήματά τους οι γεωργοί μας. Χάνουμε πολλούς νέους που φεύγουν από την Ήπεθρο και πηγαίνουν στα αστικά κέντρα. Τα, οι αναπτυξιακές δυνατότητες της γεωργίας μας έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. Η ανάπτυξη στην Ήπεθρο είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι μαζικής, ε, από ό,τι στα αστικά κέντρα και δικαία οι αγρότες μας διαμαρτύρονται. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για ανάπτυξη της υπαίθρου Αϊφόρο βιώσιμη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βάιντερ. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό, την έκθεση αυτή, γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικά κριτήρια και προϋποθέσεις για μια νέα γεωργική πολιτική. Πρέπει να έχουμε απευθείας υποστήριξη στον γεωργικό προϋπολογισμό, από τον γεωργικό προϋπολογισμό, απευθείας ενισχύσεις. Η δε πατρίδα μου η Λετωνία είναι εδώ και μερικά χρόνια βέβαια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως μόνο 90 ευρώ ανά εκτάριο από κοινοτικέ ενισχύσεις λαμβάνουν οι αγρότες μας, ενώ οι Έλληνες γεωργοί λαμβάνουν 550 ευρώ και οι Γερμανοί 300 ανά εκτάριο σε απευθεία ενισχύσεις. Αυτή είναι η αδικία, αυτό είναι το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων ή μικρών και μεγάλων κρατών μελών. Και αυτό βέβαια δεν ευνοεί την ανάπτυξη στα μικρότερα στα νέα συγγνώμη κράτη-μέλη. Χρειάζεται να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία. Δεν το Ευχαριστούμε. Ο Στάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση Λάιον και σε αρκετά σημεία. Πρέπει να ομολογήσω ότι είχα τις επιφυλάξεις μου για λόγους εθνικούς. Όμως η έκθεση Λάιον είναι καλή έκθεση. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ το στόχο της μεταρρύθμισης της κοινή πολιτικής. Όμως εγώ προερχόμενο από ένα μικρό κράτος πρέπει να πω ότι έχουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες από ό,τι φερειπίνει η Γερμανία στη γεωργία μας δεν είναι συμβατά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς στην ε, χώρα μου με αυτά τα οποία ορίζει η κοινή πολιτική. Όμως, πρέπει τα μικρά κράτη να έχουν ιδιαίτερη προστασία. Πρέπει να μεριμνήσουμε ιδιαίτερα για τα μικρότερα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δέβιτ Μάρτιν έχει το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση. Λάιον, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, πρέπει να διαχειριστούν τους προπολογισμού του Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αντιμετωπίζουν περικοπές στις αμοιβέ και τις συνταξιοδοτήσεις τους. Ε, πολλοί, οι πολλοί φυλακισμένοι επίσης απελευθερώνονται γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος των σοπανιστικών ιδρυμάτων. Το Ευρω... Στο Ευρωκοινοβούλιο οι εκπρόσωποι της Βρετανικής κυβέρνησης που είναι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές πιστεύουν ότι θα πρέπει να περιμένουν γεωργικέ δαπάνες ως το 2013 και μετά στα επίπεδα αυτού του έτους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι τελείως απαράδεκτα, απαράδεκτο μάλλον η γεωργική κοινότητα να μην λαμβάνει υπόψη το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία. Εάν το εισόδημα των υπόλοιπων πολιτών περιορίζεται, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και, στα, ε, και στο γεωργικό τομέα. Οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει λοιπόν και τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να παραμείνουν εδώ σε ένα κοινό μέτωπο, ιδάλω θα αντιμετωπίσουν το ίδιο τίμημα. Ευχαριστούμε ο κύριος Σάιτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι πολιτικοί ηθήνοντες είδαν ε, ποιε ήταν οι συνέπειε του πολέμου και γι' αυτό ήθελαν να προωθήσουν την κοινή γεωργική πολιτική και την επιστηστική ασφάλεια. Όμως αν δείτε 60 χρόνια μετά τι έγινε μετά την ε, θέσπιση της Ευρωπαϊκής Γεωργικής Πολιτικής, το συμπέρασμα είναι ότι οι πολίτες πληρώνουν τρία φορές περισσότερο για την γραφειοκρατία, για τους ε, φόρους και για το υψηλό κόστο των προϊόντων παρά για την ουσία. Θα πρέπει λοιπόν, μιλώντα για τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική, θα έπρεπε καλύτερα να μιλάμε για την πλήρη κατάργησή τη, Να την καταργήσουμε ώστε να επιτρέψουμε στου φιλελεύθερου γεωργού να ε, μπορέσουν να, ακμάσουν. Να επιτρέψουμε στους φορολογουμένου να εξοικονομήσουν τα χρήματά του. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα να αρπάξουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ευχαριστούμε. Και τώρα τελευταίος η κυρία Γιατεμάκη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Περψήφισα την έκθεση. Λάιον. Τη βρίσκω καλά ισορροπημένη. Θεωρώ ότι είναι μια έκθεση η οποία εξασφαλίζει πως σε ολόκληρη την Ευρώπη θα υπάρχει γεωργία, θα συνεχιστεί η γεωργική δραστηριότητα, η παραγωγή τροφίμων, θα εξασφαλιστεί η επιστηστική ασφάλεια. σε κάποια σημεία διαφοροποιήθηκα στην ψηφοφορία σε σχέση με την ομάδα μου, διότι θεωρώ ότι η ρύθμιση αγοράς και η παρέμβαση σε ορισμένες καταστάσεις απαιτείται και για τη διασφάλιση των τσιπιστικής ασφάλειας και για την διαφύλαξη μιας αηφόρου παραγωγής. Péter ε, äh, äh, képviselő Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση. Έχει ιδιαίτερη σημασία ποιοτική, κοινωνική, γεωργική φυσικά. Απαραίτητο είναι διαφυλαχθεί η παραγωγή των προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε τα αλλιεύματα που κινδυνεύουν από τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Επίσης υπάρχουν οικονομικοί όροι και με δεδομένο ότι κινδυνεύουν τα ελιεύματα σε πολύ μεγάλα ποστά σε ολόκληρο τον κόσμο, έως και 50% πρέπει να δώσουμε έμφαση στην υδατοκαλλιέργεια, η οποία και θέση εργασία δημιουργεί και προσθεμένη αξία υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Χάιντερ και πάλι. Ε, Ευχαριστώ. Η έκθεση καλύπτει τις ε, οικολογικές και κοινωνικές διαστάσεις αλίας. Προσπαθεί να διαφυλάξει μια οικολογική και κοινωνική αλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αναγνωρίζει την αλία στην Ευρώπη ως και ένα παράγοντα πολιτιστικό και ως ένα παράγοντα διαφύλαξης θέσεων εργασίας. Δυστυχώς όμως. Δυστυχώς η Λετωνία έχουν τόσο μικρές ποσοστώσεις και τόσο περιορισμένη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μάλλον υποχρεωμένοι να προχωρούν σε διάλυση των σκαφών τους και να εγκαταλείπουν τη δραστηριότητα. Αυτό είναι τραγικό διότι τα 550 χιλιόμετρα των ακτών μας δεν ε, αναπτύσσονται, δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και πολλές φορές ε, βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί σε απόγνωση. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Την έκθεση αυτή την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο σήμερα και απλώ ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασχολείται με τις ίδιους πολίτες της. Και αυτό είναι ισχύει και για τις αλληλευτικές κοινότητες. Λειτουργούν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, εδώ και αιώνες και έχουν επιβιώσει χάρη στην ε, αλία. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπουμε τα ίδια πρότυπα διαβίωσης αλλά και τις ίδιους κανόνες ε, προστασίας για τα προϊόντα που έρχονται από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και αυτά που εισάγουμε. Θέλουμε να προάγουμε κι άλλο την υδατοκαλλιέργεια και έτσι να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ευχαριστώ. Τελευταίος, ο κύριος Κιμάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους εδώ για την υπομονή τους και να πω ότι όταν πρώτη φορά σκέφτηκα την κοινή αλληλευτική πολιτική σκέφτηκα ότι η θάλασσα είναι περισσότερο μέρος ε, για την... Ε, ότι από το κοινή πολιτική το ΚΑΠΑ μπορεί να σημαίνει κομμουνιστική πολιτική. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι ε, τα αποθέματα όλο και λιγοστεύουν, αλλά και οι παραπονιούνται για τι ποσοστώσει και τη μείωση τη ποσοστώσεις του. Και μα ενδιαφέρει και η διατήρηση των ελληνικών αποθεμάτων. Α δούμε πώ λειτουργούν τα οικοσυστήματα στην ε, Ισλανδία ή στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί οι αλληλεί έχουν δικαιώματα διαρκή, μόνιμα δηλαδή, τα οποία μπορούν να μεταπολίσουν, να εκχωρήσουν, να τα αφήσουν στι επόμενε γενιέ. Αυτό ίσω είναι η καλύτερη απάντηση στα προβλήματά μα, γιατί είναι έχει δείξει μέχρι τώρα την επιτυχία του. Και όχι ένα σύστημα όπω αυτό τη κοινή αγροτική πολιτική που έχει αποτύχει παταγωδό στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Και εμεί ανησυχούμε ιδιαίτερω και για την φύση. Και σταματούμε εδώ για να ξαναρχίσουμε στις 3.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 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, πέραν της ε, περιπτώσεις του Φαραή Βαγκού υπάρχει η περίπτωση της εκμεταλλεύσεως των διαμαντιών. Υπάρχει η διαδικασία του Κίμπερλε και